συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε ε, στο πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας, ε, πρέπει να σας θέσω ένα θέμα διαδικαστικό. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε την Επιτροπή για Εσωτερικές Υποθέσεις και Αστικές Ελευθερίες να την παρακαλέσει να επιληφθεί της ε, κατάστασης στην Δανία λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία στη χώρα αυτή για την ε, καταβολή κοινωνικών επιδομάτων στους πρόσφυγες. Μετά λοιπόν από επιθυμία της ε, διάσκεψης των Προέδρων παρακάλεσα την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να επιληφθεί του θέματος. Οι συντονιστές της Επιτροπής ε, πλειοψηφικά αποφάσισαν το θέμα να μην το συζητήσουν πάρα αυτά, αλλά να το μεταθέσουν σε μία μεταγενέστερη συνεδρίαση. Και αυτό μου το ανακοίνασε ο κύριος Μωράς, ο πρόεδρος σε μία επιστολή. Μου το ανακοίνωσε λοιπόν ο πρόεδρος Επιτροπής σε μία επιστολή στις 15 Ιανουαρίου. Μου είπε λοιπόν, ανακοινώνει, ότι η Επιτροπή θα επιληφθεί αυτού του θέματος ε, στο τέλος Ιανουαρίου. Κατόπιν ήρθε σε επαφή μαζί μου ο κύριος Λάμπερτς με την παράκληση της πολιτικής του ομάδας να κάνουμε ό,τι μπορούμε πλειοψηφικά να προχωρήσουμε το θέμα χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Να τεθεί το θέμα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Κατόπιν τούτου ήρθα σε επαφή με όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δω κατά πόσο διαμορφώνεται πλειοψηφία ή όχι. Η αδιαμφισβήτητη λοιπόν πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων ε, μονακίνωσε σήμερα το πρωί ότι δεν θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να τεθεί στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Και αυτό έπρεπε να σας το ανακοινώσω. Ο κύριος Λάμπερτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας, Πρόεδρε. Ε, προφανώς υπάρχουν πολλοί που δεν επιθυμούν να συζητηθεί η κατάσταση στη Δανία. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για, το, για θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο η